Okay, ladies and gentlemen. Let's hope a few more of the members filter in. Αρχίζουμε κυρίες και κύριοι, ελπίζω στο μεταξύ να έρθουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους σε αυτή τη μήνυα ακρόαση για τον κανονισμό για τις λιπενικές υπηρεσίες. Η πρόσβαση στις λιμενικές υπηρεσίες και χρηματοοικονομική διαφάνεια στα λιμάνια. Έχουμε τρεις ε, ή πέντε μάλλον πολύ διακριμένους καλεσμένους, τον κύριο Ρίτσαρτ Πέρτ από το, από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Στεφάνο Μπενάλντο, Ρονάλντο είδα στην αρχή, από το λιμεναρχείο της Βενετίας, είναι τον Οργανισμό Λιμένος μάλλον Βενετίας, τον κύριο Βίκτορ Σον Μάρκες από το Ρότερνταμ. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε για τα λιμάνια στην Ευρώπη αν δεν αναφέρουμε και το Ρότερνταμ. Την κυρία Ναρίνα Μακέλη από την Ένωση Λιμένων Φιλανδίας, τον Αζαν Κλωτεριέ ε, από το Φορέα Διαχείρισης ε, του Λιμένα της Μασαλίας. Η δομή είναι κάπως διαφορετική στη σημερινή ακρόαση, γιατί θα γίνεται συζήτηση αμέσως μετά την κάθε παρουσίαση. Οπότε θα ακούμε έναν ομιλητή και μετά θα έχουμε γύρω ερωταπαντήσεων. Πρώτα θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Ρίτσαρτ. Αυτό που μου αρέσει στο Ρίτσαρτ είναι που το πρώτο ε, που μου είπε είναι ελπίζω να είσαι αυστηρός με το σφυρί. Χαίρομαι πολύ που έχω τέτοια φήμη σκληρού. Από, ε, για ένα πεντάλεπτο λοιπόν ο Ρίτσαρτ από το Ηνωμένο Βασίλειο και από τη μεγαλύτερη Ένωση Λιμένων. Σας ευχαριστώ για την διοργάνωση αυτής της δημόσιας ακρόασης και την καταπληκτική ευκαιρία που μας δίνεται να παρουσιάσουμε τη θέση των λιμένων για τον κανονισμό αυτό. Και είναι κρίμα που δεν είχαμε αρκετές διαβουλεύσεις πριν την κατάθεση της πρώτης του κανονισμού. Στο πεντάλεπτο που έχω θα ήθελα να σας ε, δώσω κάποια στοιχεία για το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί φαντάζομαι έχουμε διαφορετικό τρόπο για, να, για τον τρόπο διαχείριση των λιμένων μας. Και μετά θα αναφερθώ σε κάποιες ε, από τις ερωτήσεις ε, που θα μου υποβληθούν. Εμείς έχουμε το μεγαλύτερο τομέα λιμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 120 εμπορικά λιμάνια, 44 από αυτά ανήκουν στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, οπότε μας επηρεάζει άμεσα αυτός ε, ο κανονισμός. Και μάλιστα έχουμε και ιδιωτικούς λιμένες ή λιμένες από ιδιωτικούς ε, τομείς ή από ιδιωτική χρηματοδότηση. Και ο τρόπος που γίνεται η διαχείριση αυτών των λιμένων συνάδει και με την κυβερνητική πολιτική, γιατί όλες οι κυβερνήσεις ε, δεν ε, επιχορηγούν τα λιμάνια προκειμένου να αναπτύσσεται ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ τους. Τα λιμάνια ε, συμβάλλουν στην Βρετανική οικονομία. Το 95% του Βρετανικού Διεθνούς Εμπορίου περνάει από τα Βρετανικά λιμάνια και διευκολύνουν πολλές, πολλούς κλάδους, ιδιαίτερα τις ενέργειες. συμβάλλουν ε, στη δημιουργία θέσεων απασχόληση και αντιπροσωπεύουν περίπου το 1% του συνολικού ΑΕΠ ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Μπορεί να μην βλέπετε τις λεπτομέρειες στον κανόνα αυτό, αλλά βλέπετε ότι έχουμε πολλά ε, λιμάνια σε πολλά σημεία της χώρας με σημαντικό όγκο εργασιών και μάλιστα πολύ, πολύ κοντά, το πολύ 120 χιλιόμετρα από τα λιμάνια, έχουμε σημαντικά αστικά κέντρα. Γι' αυτό και υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των λιμανιών. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και συμβάλλει στον τρόπο ανάπτυξης ε, του τομέα αυτού. Ε, είμαστε μια, ε, ένας κλάδος που ανανεώνεται συνέχεια με πολύ ψηλό επίπεδο επενδύσεων, γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο υπολογίζεται, Επίσης έχουμε πολύ σημαντική παραγωγικότητα, 40% πάνω από τον μέσο όρο του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε εξαιρετικές βιομηχανικές σχέσεις στα λιμάνια, ενισχυμένη ασφάλεια και περιβαλλοντικές επιδόσεις. Επίσης έχουμε πολύ καλές διασυνδέσεις με την εδωχώρα, οδικές, σιδηροδρομικές και μεσοτερικές πλωτές οδούς. Οπότε ε, το 2010 διαπιστώσαμε από τον αρμόδιο φορέα ότι και ο, κανονισμό, ο ανταγωνισμός λειτουργεί πολύ καλά στα Βρετανικά λιμάνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο κανονισμό, ε, είμαστε υπέρ των αρχών ε, της κάλυψης των προβλημάτων της αγοράς, της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της βελτίωσης της παραγωγικότητας. Πολύ φοβόμαστε όμως ότι ο κανονισμός αυτός θα επέμβει και σε τομεί που η αγορά λειτουργεί εύρυθμα. Για παράδειγμα, το κεφάλαιο 2 θα δημιουργήσει γραφειοκρατία επιπλέον κόστο και θα έρθει σε αντίφαση με κανονιστικέ, ε, συμβατικές και εργασιακές δομές. Και μάλιστα θα δημιουργηθεί έλλειψη ασφάλειας εκεί που γίνεται αυτοδιαχείριση από τα λιμάνια. Έχουμε το κεφάλαιο 3 για τις χρηματοοικονομικές διατάξεις και τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, γιατί τα λιμάνια δεν θα μπορούν πια να ε, έχουν εμπορικέ δραστηριότητες ε, και επίση είναι σαφή και ο μελλοντικός ρόλος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά τη χρέωση, κάτι που δημιουργεί αβεβαιότητα και δημιουργείται και ένα νέο επίπεδο γραφειοκρατίας εξαιτία ε, του φορέα, του νέου φορέα που προτείνεται. Θέλουμε λοιπόν τον εξάρτητο υποπτικό φορέα. Θέλουμε σίγουρα αποτελεσματικότητα, αλλά όχι να δημιουργηθεί ένας ασφικτικός κλειός με τις νέες διατάξεις, κάτι που θα επιτείνει την, ε, την αβεβαιότητα και θα είναι δύσκολο να προσελκύσει και επενδύσεις. Οπότε θα ήθελα να διακοπούν οι συζητήσεις για τον κανονισμό προκειμένου να, ε, να αποτιμηθεί δεόντως ο αντίκτυπος ε, των νέων κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες και το πρόβλημα της πρωτοβουλίες για τις κρατικές ενισχύσεις. Ε, δεν θα πρέπει οι προτάσεις αυτές να αναχαιτήσουν τη δραστηριότητα των Βρετανικών λιμανιών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις που μας έστειλε ο εισηγητής. Ακροθυγή απάντηση. Καταρχήν, ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού και την πρόσβαση στην αγορά. Δεν θεωρούμε ότι οι διατάξει για την πρόσβαση στην αγορά αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί τα λιμάνια μα είναι εμπορικά Τώρα, σε ό,τι αφορά τον εχώριο ε, πάροχο του άρθρου 9, είναι υπερβολικά περιοριστικός ο ορισμός, ε, ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά την υποχρέωση της παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Σε ό,τι αφορά τα τέλη, δεν είναι πολύ ισορροπημένος ο κανονισμός, γιατί σε μια ανταγωνιστική αγορά θα πρέπει να ισχύουν οι κανονικές συνθήκες για τη χρέωση και τα τέλη. Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά λιμάνια, ιδιαίτερο θέμα για το Ηνωμένο Βασίλειο, θέλουμε ενδεχομένως να υπαχθούμε σε κάποια εξαίρεση από τον κανονισμό. Πάντως ε, θα προτιμούσαμε να αποσυρθεί τελείως η πρόταση κανονισμού, να γίνει ενδελεχής και εκτενή συζήτηση και μετά να ξαναρχίσουμε. Σε ό,τι αφορά τον εποπτικό φορέα, τον ανεξάρτητο εποπτικό φορέα, εμείς με το ε, γραφείο που έχουμε για τον θεμητό ανταγωνισμό και και την Επιτροπή Ανταγωνισμού θεωρούμε ότι υπάρχει κατάλληλη εποπτεία. Δεν χρειαζόμαστε έναν επιπλέον ανεξάρτητο εποπτικό φορέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα κάνω εγώ τις πρώτες ερωτήσεις. Θα ξεκινήσουμε τους ομιλητές, μετά θα κάνω εγώ κάποιες ερωτήσεις και μετά οι βουλευτές. Κύριε Φλέκενστάιν, έχετε κάποια ερώτηση λοιπόν για τον κύριο Μπέρντ. Όχι, όχι ακόμα, ωραία. Κάποιος άλλος έχει ερωτήσεις. Ε, μπορείτε να κάνετε και παρατήρηση αν θέλετε, όχι μόνο ερώτηση. Μάλιστα, σύντομα. Όσον αφορά τα ιδιωτικά λιμάνια, πρέπει νομίζω να διακρίνουμε, ειδικά όσον αφορά το καθεστώς τους, μεταξύ αυτά στα οποία παίζει ρόλο το δημόσιο χρήμα και στα καθαρά ιδιωτικά. Δεύτερον, που πρέπει να σκεφτούμε είναι το μονοπόλιο το οποίο ε, για το χρήστη είναι κάτι το άσχημο. Και βέβαια του είναι διάφορα αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το μονοπόλιο. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να ληφθούν υπόψη αυτά. Μάλιστα. Κύριος Κούν, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να μάθω τι γίνεται με τους πλοηγούς στα λιμάνια του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι δημόσια υπηρεσία ή ιδιωτική. Ε, ανεφοδιασμός, ρημουλκά, όλα αυτά. Υπάρχει επίσης κάποιος διαχωρισμός δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων ή έχουμε κάποια μορφή συνεργασίας με ΕΣΔΙΤ ε, ή έχουμε δηλαδή ιδιωτικά λιμάνια με κάποιες δημόσιες επενδύσεις. Σας ευχαριστώ κύριος Μπράντμπορν. Ευχαριστώ Μπράιν. Μια απλή ερώτηση έχω. Νομίζω ο, ο κύριος Μπέρν ε, αναφέρθηκε σε μια διαφάνεια. Έχω δίκαιο ότι ανεξαρτήτως των προτάσεων της οδηγίας αυτής τα λιμάνια στο Ρωμαίο Βασίλειο υπόκειται στους ε, κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ανταγωνισμού. Κάποιος άλλος? Όχι. Εγώ λοιπόν, λέει ο η δική μου ερώτηση μιλήσατε για τα ιδιωτικά λιμάνια και την οικονομική διαφάνεια. Τα λιμάνια του Ιρμού Βασιλείου έχουν κάποιο πρόβλημα με τις προτάσεις οικονομικής ε, διαφάνειας ε, σας δυσκολεύουν σας δυσκολεύει π.χ. το να ξέρουν οι ανταγωνιστές σας το τι χρεώνεται για το χ και το ψ και πριν φύγει εδώ πέρα η κυρία με το τσάι. Ε, καφέ, τι να κάνουμε άμα δεν έχει. Ελ τι να κάνουμε. Ξέχασα το, το τσάι μου και λίγο γάλα σας παρακαλώ. Η δεύτερη ερώτηση. Στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα είπατε πως θεωρείτε πως πρέπει να απορριφθεί εντελώς η πρόταση αυτή. Μπορείτε να μας εξηγήσετε το, το γιατί. Γιατί θέλετε να ακολουθήσουμε τη λεγόμενη πυρηνική επιλογή. Καλό βεβαίως, αλλά εκεί πέρα η από εκεί πλευρά θα πάθει εγκεφαλικό. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν γιατί θεωρείτε πως πρέπει να απορριφθεί η πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πολλά με έχουν πει, αλλά ε, τι να σου πω. Για πυρηνικά πρώτη φορά το ακούω. Λοιπόν, με τη σειρά. Ο κύριος ε, Φλάγκενστάιν ε, έκανε μια καλή διάκριση μεταξύ ε, λιπανιών που είναι εντελώς ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα και κάποια μικτής χρηματοδότησης. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ιδιωτική χρηματοδότηση. Ελάχιστα είναι τα δημόσια κονδύλια για συγκεκριμένους στόχους, ουσιαστικά περιβαλλοντικούς για να ενθαρρυνθεί δηλαδή η μεταφορά διαθαλάσσης και περιφερειακή χρηματοδότηση. Αλλά η καθημερινή λειτουργία χρηματοδοτείται ιδιωτικά. Και, σωστό αυτό. Και πολύ καλή ερώτηση για τα μονοπόλια. Γιατί αν κάποιος έχει μονοπωλιακή θέση, εάν είναι είτε είναι δημόσια είτε ιδιωτική χρηματοδότηση υπάρχουν ζητήματα. Νομίζω όμως σας έδειξα πως σε γενικές γραμμές στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε μια δομή η οποία επιτρέπει τον ανταγωνισμό. Και αυτή ήταν οπωσδήποτε η άποψη των αρχών ανταγωνισμού όταν εξέτασαν την κατάσταση πριν από δύο χρόνια, κάνα δύο χρόνια. Βεβαίω, στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν ζητήματα κάποιων μεμονωμένων μονοπωλίων, είναι θέμα των αρχών ανταγωνισμού και αν υπάρξει κάποια καταγγελία θα διαρευνηθεί. Ο κύριος Κούν ρώτησε για το τι γίνεται με τους πλοηγούς. Κατά κανόνα είναι, ανήκουν και είναι υπάλληλοι του λιμενός. Είτε ε, με ανάθεση είτε υπάλληλοι του λιμένος. Αυτά τα δύο υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάποια εταιρεία δηλαδή η οποία έρχεται και προσφέρει τις υπηρεσίες. Οι πλοηγοί ανησυχούν επίσης για την πρόταση αυτή και δεν είναι οι μόνοι. Και οπωσδήποτε και άλλοι θα ανησυχούν. Ελπίζω να απάντησα και στην άλλη σας ερώτηση. Κύριε Φλέκενστάιν, η ερώτηση του κυρίου Μπραντμπον. Πράγματι, ισχύει το Γενικό Δίκαιο του Ανταγωνισμού της Ένωσης ε, και οι διατάξεις περί δημοσίων προμηθειών. Οπότε η οδηγία για συμβάσεις παραχώρησης που μόλις πέρασε θα ισχύσει για τους λιμένες ε, εκείνους όπου η σύμβαση παραχώρησης είναι πάνω από το ελάχιστο όριο. Και εδώ πέρα ανησυχούμε ακριβώς γιατί υπάρχει πιθανότητα σοβαρών αλλαγών, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικώ. Η οδηγία αυτή δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ε, και θα έχει σοβαρό αντίκτυπο και ε, ξέρω πως και εμείς και πολλοί συνάδελφοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσουν προσεκτικά τις πιθανές συνέπειες πριν ε, προτείνουν κάποιο τρόπο να να ρυθμιστούν οι υπηρεσίες, γιατί και οι υπηρεσίες θα καλύπτονται από την οδηγία περί συμβάσεων παραχώρησης. Κύριε Πρόεδρε, οι δικέ σας οι ερωτήσεις για την διαφάνεια. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό μας προξενεί τις λιγότερες δυσκολίες, αλλά είναι μια αρχή που υπάρχει ήδη στο ευρωπαϊκό δίκαιο με την οδηγία περί διαφάνειας και προφανώς οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν εθνικές και διεθνείς ε, προδιαγραφές. Π.χ. αν γίνεται κάτι για τις ε, κρατικές ενισχύσεις πρέπει να υπάρχουν κάποιες σχετικές διατάξεις. Οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να δούμε ε, και στο μέλλον σε οποιαδήποτε επαναξέταση του κανονισμού. Και το τελευταίο ερώτημα περί απόρριψης. Εμείς θα προτιμούσαμε να αποσυρθεί και να επανεποβληθεί ο κανονισμός. Γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία αν συζητηθούν με τρόπο ανοιχτό και φιλικό και επικοδομητικό και έχουμε σχετικά θετική εμπειρία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε πως ε, θα επιληθούν με τρόπο λογικό και θα έτσι θα αντιμετωπιστεί η τεράστια ποικιλία ε, λιμανιών που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το ακούσετε και από τους άλλους ομιλητές. Είναι ατυχές το ότι έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που είναι ζουρλομανδίας όπως τη χαρακτήρισε η ΕΣΠΟ. Αυτά λοιπόν, από εκεί η πρότασή μας. Μάλιστα. Κοιτάξτε, καθυστερούμε λίγο, οπότε κνούτ λίγο σύντομα. Ένα θέμα μόνο, στο οποίο νομίζω συμφωνούν όλοι. Μπορούμε να μιλάμε για τα κριτήρια διαφάνειας των τιμών. Αλλά βεβαίως και ο ανταγωνισμός μεταξύ λιμανιών πρέπει να είναι δυνατός. Να υπάρχει δυνατότητα ελκυστικών προσφορών, να προσελκύσει δηλαδή κάποιος γραμμές σε άλλο λιμάνι. Αλλιώς θα ήταν αντικείμενο συνεννόησης και όχι ανταγωνισμού. Δεν νομίζω να είναι αυτό το αντικείμενο της οδηγίας. Μάλιστα δεν ξέρω αν θα θέλατε να απαντήσετε. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Δυστυχώς το κεφάλαιο 3 του κανονισμού παρεμβαίνει με την κανονική αυτή εμπορική λειτουργία που έχει τεράστια σημασία. Ναι, βεβαίω. Σας ευχαριστούμε. Βενετία. Κατόπιν. Βεβαίως ο Πάολο έπρεπε να είναι εδώ. Δυστυχώς δεν είναι εδώ. Αλλά ήθελα να κάνω πολύ πιο όμορφο στη θέση του. Ε, τον Στέφανο Μπενάλντο από την, ε, τον Οργανισμό Λιμένος Βενετίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα είμαι τόσο καλός όσο ο μιλητής που προηγήθηκε, ούτε θα σας πω τις λεπτομέρειες του Ιταλικού λιμενικού συστήματος. Θα προσπαθήσω να περάσω απευθείας στα σημεία που αφορούν τη σημερινή συζήτηση και πρόσκληση η πρόταση κανονισμού για τις λιμενικές υπηρεσίες και η δημοσιονομική της προκοδότηση. Εδώ, από τη δική μας τουλάχιστον τη Σκοπιά, το θέμα αυτό, το όλο ζήτημα, δεν μπορεί να εξεταστεί εάν δεν πούμε δύο λόγια για το τοπίο εντός το οποίο εντάσσεται αυτό το ζήτημα, αυτό το θέμα συζήτησης. Έχει να κάνει με την οικονομική λοιπόν, με το οικονομικό σκέλος και το νομοθετικό, το νομικό σκέλος. Από τη σκοπιά της οικονομίας είναι σαφές. Δεν μπορεί κανείς να αντικρούσει ότι το σημερινό λιμενικό και θαλάσσιο σύστημα, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, περνά δύο μεγάλες αλλαγές, δύο μεγάλα φαινόμενα. Ο γιγαντισμός, θα έλεγα, των λιμανιών από τη μια πλευρά, διότι οι εφοπλιστικές εταιρείες κάνουν ό,τι μπορούν για να αξιοποιήσουν τις οικονομικές δυνατότητες και κατά τα άλλα η εξάπλωση των αγορών και η προστασία των λιμένων προκειμένου να αυξήσει κανείς τον ανταγωνισμό μεταξύ των λιμένων. Μία, έναν ανταγωνισμό που μέχρι, μέχρι μερικά χρόνια πριν ήταν ανταγωνισμός των τέρμιναλ μέσα στα ίδια τα λιμάνια. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να είμαστε εύστοχοι στην παρέμβαση μας, ιδέως προς τη νομική πλευρά του θέματος, δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει ότι ο κανονισμός αυτός, η πρόταση αυτή κανονισμού, έχει να κάνει με το όλο νομικό πλαίσιο που προκύπτει από τη συνθήκη του 1957 που ορίζει την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Μία κοινότητα υπό την πλήρη νομική έννοια. Οι στόχοι τώρα οι στόχοι που μας αφορούν από την πρόταση κανονισμού είναι η δημιουργία της έννοιας του Common Level Playing Field, ή ίσοι κανόνες ε, ανταγωνισμού και παιχνιδιού, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε. Και θα πρέπει να το δούμε από την κοινοτική, την ε, ενωσιακή ε, σκοπιά. Ως προς τους στόχους λοιπόν του ίδιου του κανονισμού, να σας δώσω το παράδειγμα της Ιταλίας. Η κατάσταση συνοπτικά περιγράφεται σε αυτόν τον πίνακα, σε αυτό το διάγραμμα. Σε ό,τι αφορά τις χερσαίες και λιμενικές υπηρεσίες και στις διάφορες ε, οριζόντιες γραμμές, την διαφορά κυβερνητική Euro Imperi και την αγορέα την Euro Gestionis, βλέπουμε ότι στην Ιταλική τουλάχιστον ε, περίπτωση, είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα, εντάσσονται στο κουτάκι το κάπως πιο κόκκινο που βλέπετε στο, στη διαφάνεια. Έχουν να κάνουν με την λιμενική αρχή και το λιμενικό φορέα που όμως είναι πολύ ε, αδύναμος. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο κανονισμός που προτίθηκε και θα ψηφιστεί θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα να διευρυνθεί το πεδίο δράσης και αρμοδιότητας των λιμενικών αρχών. η αρχή δηλαδή που διαχειρίζεται τον λιμένα προκειμένου να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες ε, διακυβέρνησης governance και να μπορέσει να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα ενός λιμένα. Ό,τι αφορά τις υπηρεσίες που θα πρέπει να ενταχθούν εδώ, ένα ερώτημα που τέθηκε και προηγουμένω, οι υπηρεσίε θα πρέπει να καλύπτονται από τον κανονισμό. Εμεί θεωρούμε ότι όλε οι υπηρεσίε πρέπει να καλύπτονται από την γραμμή TFEU, την Συνθήκη Λειτουργίας δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους γενικούς κανόνες που προκύπτουν από αυτή. Δεν θα πρέπει να υπάρχει εξαίρεση κατά την άποψή μας. Η γενική ιδέα τώρα που θεωρούμε ότι είναι σωστή μέσα στον κανονισμό είναι να υπάρξει ένα ορισμό σε κοινοτικό επίπεδο από την πλευρά των θεσμικών οργάνων ω προ ένα γενικό πλαίσιο κοινών κανόνων, στι οποίε θα συμφωνούν όλοι και οι οποίε μετά θα επεξηγούνται ανάλογα με τι εθνικέ ιδιαιτερότητε και ανάγκε και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν διεθνεί κανόνε, κοινοτικοί, αλλά μετά και προσαρμογή στι ε, τοπικέ και περιφερειακέ ανάγκε. Εδώ θα μπορούσε να μα εξυπηρετήσει στην περίπτωσή μα και καθώ μιλάω για την Ιταλία ούτω ή άλλω, τα 4-5 σημεία τα οποία παριθμώνται εδώ στην διαφάνεια. Δηλαδή, να αποφύγουμε ως τώρα τη διάκριση μεταξύ των ε, θαλάσσιων ε, λιμενικών αρχών και των αρχών που προκύπτουν από τις υποδομές, θα πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός πολύ σαφέστερος. Ε, δεν απηχείται όμως η πρόταση, δεν αντικατοπτρίζεται την Ιταλική πραγματικότητα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ώρα. Το τι θα γίνεται λόγω χάρη με του επιβάτε όταν είναι φορτίο, με συγχωρείτε για τον όρο, μπορεί να σα ακουστεί κάπως τολμηρό, αλλά στην Ιταλία δεν ε, υπόκειται σε δασμολόγηση όπω τα εμπορεύματα, τα υπόλοιπα φορτία. Το πιο σημαντικό εδώ, επειδή το λέγαμε πριν και μιλήσαμε για διαφάνεια στι τιμέ, διαφάνεια στους δασμού που επιβάλλονται, και το τι trade-off θα υπάρχει, τι αντάλλαγμα με την ανταγωνιστικότητα. Σε ό,τι μα αφορά λοιπόν, το σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι τιμές, οι ταρίφες ορίζονται σε μια βάση εθελοντική, διαφορετικά από το σύστημα που εφαρμόζεται αλλού τώρα. Συνεχίζω με κάτι που νομίζω ότι δεν ε, είναι στην ίδια λογική με τους υπόλοιπους συζητητές, κάτι που θεωρώ σημαντικό πρόεδρε, ο ρόλος της υποπτικής αρχής. Για μας είναι απαραίτητο αυτό απαραίτητο μέσα σε μια λογική του common level playing field για να υπάρχει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στα θαλάσσια ζητήματα και όχι εθνικός κατακαιρματισμός. Όχι, θα πρέπει να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Γενική Αρχή με ε, υποδιέρεση σε εθνικά επίπεδα και μετά ε, με προσαρμογή στο τοπικό ε, επίπεδο. Βλέπετε τι γίνεται λόγω χάρη με, την Αμερικα... με τον Αμερικανικό φορέα, την ε, Ομοσπονδιακή Επιτροπή για τα Θελάσσια Ζητήματα, που είναι ένας φορέας υπεύθυνο να ρυθμίζει το σύστημα μεταφοράς διεθνώς της Θελάσσιας οδούς και βεβαίως τις εισαγωγές και εξηγωγές. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, κλείνω. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις προς τον κύριο Μπενάλντο, παρακαλώ. Ο κύριος Φλάκενστάιν. Μια ερώτηση. Μόνο το μιλήσετε για αυτούς τους συμβουλευτικούς φορείς που λέτε πως δεν πρέπει να είναι εθνική αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το ερώτημά μου είναι μέχρι τώρα η εφαρμογή του κανονισμού από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη ε, εφαρμόζεται δηλαδή από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη και επιτηρείται από αυτούς. Γιατί χρειάζεται για αυτό το ζήτημα ε, εποπτικός ε, φορέας. Εντάξει, για παράπονα και τα λοιπά το καταλαβαίνω. Αλλά για το άλλο κομμάτι θεωρώ πως είναι περιττή η ύπαρξή του. Υπάρχουν τα κράτη-μέλη, υπάρχει η Κομισιόν. Ε, δεν είναι δυνατόν, δεν έχει ξαναδημιουργηθεί δηλαδή φορέας για να ασχολείται με έναν μόνο κανονισμό. Κύριε Μπραντών. Ευχαριστώ. Αν σας κατάλαβα καλά, είπατε σε, μιλήσατε για ανταγωνισμό, για διαχείριση του ανταγωνισμού. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Διαχείριση του ανταγωνισμού προσπάθησα να παρακολουθήσω και από τις διαφάνειες. Ουσιαστικά θέλετε έναν κανονιστικό έλεγχο της ε, διαδικασίας του ανταγωνισμού. Γιατί κατά τη γνώμη μου όταν έχουμε ανταγωνισμό, έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ ε, είτε μονομένων λιμένων της ίδιας χώρας, είτε μεταξύ λιμένων σε διαφορετικές χώρες. Τι εννοείται με τη διαχείριση του ανταγωνισμού, γιατί ο ανταγωνισμός ε, δράζεται στην αγορά. Δεν εννοείται διαχείριση του ανταγωνισμού, κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, είστε ευχαριστημένος σε γενικές γραμμές με την πρόταση. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ποια κριτική θα ασκούσατε και τι σας ανησυχεί εσάς. Πρώτον, επειδή είπατε πως είναι καλό να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό εποπτικό όργανο όπως η Αμερικανική Επιτροπή Ναυτιλίας θεωρείται πως θα πρέπει να εξετάζει γενικώ την ε, θαλάσσια πολιτική πέρα από τα λιμάνια. Δεν ξέρω τι, τι κάνετε εσείς. Εμείς από το Βαμβούργο που είμαι τα κάνουμε κάπως διαφορετικά. Θα ήθελα και εγώ, Στέφανο, να κάνω μια ερώτηση. Συνεχίζοντας κατά κάποιο τρόπο το συλλογισμό του κ. Μπράτμπερν. θεωρείτε ότι η πρόταση δεν είναι αρκετά φιλόδοξη. Πιστεύετε ότι και η διακίνηση φορτίου θα πρέπει να εντάσσεται στο πακέτο για τις λιμενικές υπηρεσίες. Γιατί για αυτό το σημείο υπάρχει αντιπαράθεση. Είτε είναι κανείς υπέρ της ένταξης της διακίνησης φορτίου στον κανονισμό, είτε ε, κατά. Γιατί έχουμε ένα πακέτο για τις λιμενικές υπηρεσίες, από το οποίο όμως ε, εξαιρούνται πολλά πράγματα. Και εδώ έχουμε διάσταση απόψεων, έχουμε δύο-τρία στρατόπεδα για τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω όμως εσείς ε, τι ακριβώς πιστεύετε. Συμφωνείτε ε, με την εξαίρεση της διακίνησης φορτίου και κάποιων άλλων θεμάτων από τον κανονισμό ή θεωρείτε ότι πρέπει να ε, επαναφέρουμε στον κανονισμό. Κύριο κύριος Κουμουτσάκος έχει το λόγο. δύο ερωτήσεις πρώτη, αν θεωρείτε ότι ο καινούριο κανονισμός, ο υποσυζήτηση... Is there a translation? Do you have a translation from Greek to... Yeah, okay. Yes. Okay. So, uh, η, η πρώτη ερώτηση είναι αν uh, κατά τη γνώμη σας... Okay now? Okay. Once again. Το πρώτο ερώτημα είναι αν πιστεύετε ότι ο κανονισμός δημιουργεί διοικητικές επιπλοκές. Περισσότερο από διοικητικές, θα το έλεγα, προκλήσεις ε, όπως είχαμε στο παρελθόν με την ελληνική μας πολιτική. Ποια είναι η άποψή από αυτού. Ο κανονισμός αυτός αυξάνει ή περιορίζει, ελαφραίνει το διοικητικό άχθος των αρχών και διαδικασιών. Τώρα ελπίζω να έχετε διερμηνία στα ελληνικά, από τα ελληνικά. Είναι αν... και η δεύτερη ερώτηση είναι αν ε, με τον νέο κανονισμό πιστεύετε ότι πραγματικά προετοιμάζονται τα ευρωπαϊκά λιμάνια στο να διαχειριστούν με πιο επιτυχή τρόπο το φαινόμενο της μεγέθυνσης του γιγαντισμού των πλοίων, των πλοίων και την ανάγκη να γίνεται μια σωστή διαχείριση των νέων συνθήκων, του μεγαλύτερου φορτίου και των μεγαλύτερων πλοίων. Ευχαριστώ πολύ. Στέφανο, αν ήθελες να απαντήσεις όσο το δυνατόν συντομότερα. Eh, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά, ακόμα και αν κάποιες επικαλύπτονται. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τις συγκεντρώσω. Σε ό,τι αφορά το managing body, το φορέα διαχείρισης. Καταλαβαίνω ότι ίσως δεν το εξήγησα αρκετά. Το ζήτημα είναι το εξής, πώς να το πω. Για να φτάσω και στην ερώτηση του κυρίου Φλανκεστέν. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε εθνική χώρα ρυθμίζει ανεξαρτήτως, ας πούμε, το ζήτημα. Τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό ή το εμπόριο. Αλλά για ένα θέμα τόσο ετερογενές ως προς την υλοποίηση από, των κανόνων από τις διαφορετικές χώρες, η ίδια χώρα που διαχειρίζεται και μπαίνει στην ουσία της υλοποίησης ενός κανονισμού. βάσει των δικών της ιωθώτων, της δικής της παράδοσης, αυτό μπορεί να προκαλέσει αποκλήσει, διαφορές σε σχέση με το πώ υλοποιούνται τα ίδια από σε μια άλλη χώρα. Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι πιο στραμμένες προς την αγορά, λόγω χάρη τη Νότιας Ευρώπης λιγότερο. ως προς τη δομή του ίδιου κανονισμού. ως προς τη δομή των ίδιων των λιμένων. Ε, ε, η ίδια λοιπόν υλοποίηση του ίδιου κανονισμού σε δύο διαφορετικέ χώρε μπορεί να καταλήξει σε διαφορετικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση όμω, να δώσω ένα παράδειγμα, που υπάρξει διαφορά μεταξύ υλοποίηση κανονισμού μεταξύ δύο χωρών γειτονικών, όμορων, με παρόμοια συστήματα διαχείριση, α πούμε, η Ιταλία ε, έχει γειτονικέ χώρε με τι οποίε έχει τελείω διαφορετικό σύστημα διαχείριση. Ποιο θα ορίσει ποιο σύστημα πρέπει να υπερέχει. Ε, αυτό του χώρα Α ή τη χώρα Β. Κατά την άποψή μα, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ένα φορέα διαχείριση. Ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Όχι γραφειοκρατικά όμω να δημιουργηθεί μια ακόμα υπηρεσία. Δυνατότητα να υπάρχει όμω σε επίπεδο ελέγχου κοινό, να αναφερθούν μάλλον όλα ε, αυτά σε επίπεδο ελέγχου κοινό. Για όλα αυτά τα ζητήματα. Διότι το θέμα θα συζητιέται πάντοτε μεταξύ δύο-τριών χωρών με διαφορετικέ πρακτικέ. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει διέξοδο εφόσον προκύψει διαφωνία σε τέτοιε περιπτώσει. Ελπίζω ότι απήντησα τρόπον πεινά και στις σχετικέ ερωτήσεις για το managing body των φορέων διαχείριση. Ω προ για το πώ θα χειριστούμε τον ανταγωνισμό στην αγορά. Το πρόβλημα προκύπτει από το εξή δεδομένο είναι προτεραιότητα, νομίζω μπορώ να το πω, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργανών και στο πώς έχουν καθορίσει ως τώρα την πολιτική τους, όχι για να πιέσουν την αγορά, να την εξοφίσουν κάπου, αλλά να δώσουν μια μορφή στην οικονομική ε, οικοδόμηση της Ευρώπης και προσπαθώντας να εξισορροπήσουν την ε, οικονομική ανάπτυξη που προκύπτει πολιτική και τον βιομηχανικό σχεδιασμό. Το να υπάρξει μια ρυθμιστική προσέγγιση με μια μορφή ελέγχου που να βγαίνει από την αυστηρή αντίληψη της αγοράς μας οδηγεί στο εξή. Στον τομέα της θάλασσας υπάρχουν ε, φραγμοί ε, ως προς την είσοδο. Ε, απαιτούνται υποδομές λιμένες που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα, διότι είναι πολύ μικροί λόγου χάρη, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Απο, αποκλεισμός λοιπόν από την αγορά κάποιων ε, λιμένων ε, προς όφελος άλλων. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Και σε σχέση με την τελευταία ερώτηση που έγινε από τον Πρόεδρο, αυτό που πιστεύω Εάν με ρωτούσατε τι πρέπει να γίνει με το handling, αν πρέπει να καλύπτεται ή όχι, θα έλεγα ως προς την αρχή, αυτή είναι η προσέγγιση μας, ε, όλες οι υπηρεσίες πρέπει να καλύπτονται από τις κατευθυντήριες γραμμές, με συγχωρείτε, ε, τις ε, συνθήκες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό επί της αρχής δεν είναι δίκαιο, γιατί δεν θα πρέπει να αποκλείονται κάποιες υπεράλλων και αντιστρόφως. Δεν πρέπει κάποιε υπηρεσίε να προτιμηθούν σε σχέση με κάποιε άλλε και να καλυφθούν προκειμένου να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο σκοπό. Για τι τελευταίε ερωτήσει που μου έγιναν. για το αν θα δημιουργηθεί περι, περιττέρω Δεν θα προκύψει κόστος, ή, το πώς θα διαχειριστούμε το κόστος από τον κανονισμό αυτό. Δεν το προκαλεί ο κανονισμός αυτός καθεαυτός. Η εποπτική αρχή λοιπόν του supervisory body δεν θα πρέπει να γίνει αντιληπτός κάτι που επιβαρύνει τη διοικητική δομή, το σύστημα σε ορισμένους λιμένες. σε κάποια λιμάνια λειτουργεί πάρα πολύ καλά αλλά εφόσον δημιουργούμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα, πρέπει να βγούμε από την εθνική πρόπτικη για να κρίνουμε το σύστημα αυτό και να δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι ε, αποτελέσματα θα υπήρχαν. Τι επιπτώσει. Οι Άγγλοι λόγου χάρη μπορεί να μα έλεγαν Εμά δεν μα κάνει. Οι Ολλανδοί το ίδιο, γιατί ήδη λειτουργούν πάρα πολύ καλά τα λιμάνια μα. Σε άλλε χώρε, με άλλη πραγματικότητα, μπορεί να υπήρχε ανάγκη να υπάρξει βελτίωση. Βελτίωση στη διαχείριση του ίδιου συστήματο. Και ομογενοποίηση, προκειμένου να έχουμε ανταγωνισμό στην πράξη, όχι μόνο ανταγωνισμό στην αγορά. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Μπενάλντο. Περνάμε τώρα στο λιμένο του Ρότερνταμ. Το κύριο Βίκτορ Σόνεμέκερ. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Well, thank you, Chair. I will... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με μια σύντομη παρουσίαση του λιμάνιου του Ρότερνταμ. Όλοι ξέρετε πως είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό λιμάνι. Έχουμε ένα τζίρο, μια διακίνηση 450 εκατομμυρίων τόνων ε, το χρόνο, μακράν το μεγαλύτερο λιμάνι στην ε, Ευρώπη. Είμαστε λιμάνι παγκοσμίου μεγέθους, ε, σημαντικό για την Ολλανδική και την Ευρωπαϊκή οικονομία. Και κάτι το οποίο θα ήθελα να πω είναι πως η ρύθμιση του κλάδου όπως ε, προτείνεται είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε πάρα πολύ προσεκτικά γιατί είναι κάτι το σημαντικό, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί τον μπλέκει κανείς λοιπόν σε αυτήν την υπόθεση χωρίς να ξέρει πώς ακριβώς λειτουργεί μπορεί να είναι επικίνδυνο. Η δεύτερη διαφάνεια αφορά και πάλι την δική μας τη θέση ως οργανισμού λιμένος. Έχουμε ευθύνη βεβαίως και περιβαλλοντική και κοινωνική για την ενσωμάτωση στο άμεσο περιβάλλον του λιμανιού. Πριν από δύο εβδομάδες στο Ταλίν τα λιμάνια ορίστηκαν ως πυλώνες ανάπτυξης, συμφωνώ πλήρως, στο Ρότερνταμ έχουμε μία προσέγγιση η οποία ε, καθορίζεται με βάση ένα επιχειρηματικό σχέδιο κατά το οποίο σημαίνει πως προσπαθήσαμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη της οικονομίας χωρίς δημόσια χρηματοδότηση. Και έρχομαι εδώ πέρα σε ένα από τα ε, σημαντικότερα ζητήματα, τους ίσους όρους ανταγωνισμού. Για ε, μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει νομίζω μια ανάπτυξη αυτού του θέματος στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για να ε, απαλλαγούμε από τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες πραγματικά στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των λιμανιών. Πιο συγκεκριμένα για τον κανονισμό όταν εφαρμοστεί το άρθρο αυτό περί διαφάνειας ε, θα έχουμε μια ελπίδα για να ξεκαθαρίσουμε το πώς ε, γίνονται οι κρατικές ενισχύσεις στην Ευρώπη για να έχουμε ίσως ανταγωνισμό. Δεν πρέπει κατά την απόψή μας να εξαιρεθούν τα ιδιωτικά λιμάνια από τον κανονισμό για να απαντήσω στον εισηγητή γιατί όταν λέμε ίσως όρους ανταγωνισμού αυτό σημαίνει και η ίδιο, η ίδια νομική αντιμετώπιση, όχι η διαφορετική αντιμετώπιση για διαφορετικά λιμάνια. Και αναφέρθηκε πάλι, μην ξεχνάμε, την τεράστια δύναμη της ναυτιλίας. Είδαμε προσφάτως την ε, συμμαχία των τριών μεγάλων ε, ναυτιλιακών γραμμών. Φανταστείτε να είστε ένα λιμάνι όπου βεβαίως ε, τα στοιχεία βρίσκονται δεσμευμένα σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο το οποίο δεν μετακινείται σε αντίθεση με τα απλία τότε προσπαθούμε και εμείς να το αποκριθούμε και υπάρχουν ε, από την άλλη μεριά μεγάλες δυνάμεις ε, από τη μεριά της ναυτιλίας. Βεβαίω. Συνοψίζοντας, ε, θέλουμε και εμείς να σεβαστούμε τους κανόνες της ε, συνθήκης, αλλά δεν θέλουμε να έχουμε ένα περιγραφικό σύστημα, δηλαδή δεν θέλουμε να δούμε κάποιον ε, άλλο φορέα. Υπάρχει δίκαιο του ανταγωνισμού στην Ολλανδία, λειτουργεί, έχουμε και μια διαδικασία διαβούλευσης με τους πελάτες μας και υπάρχουν ε, συστήματα στην περίπτωση κάποιας σύγκρουσης ή διαφωνίας. Έρχομαι τώρα στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Εμείς είμαστε υπέρ της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, γιατί πιστεύουμε στον ανταγωνισμό και αν για οποιονδήποτε, οποιονδήποτε λόγο γίνει κάποια επιλογή, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Νομίζω είναι σαφές αυτό και λογικό. Συγκεκριμένα για τις χρεώσεις ε, των υποδομών και πώς γίνεται αυτή η διαδικασία στο Ρότερνταμ. Είπαμε πως έχουμε μια επιχειρηματική αντιμετώπιση. Είμαστε σε συνεχή συνεννόηση με τους πελάτες μας, τους χρήστες. Ε, υπάρχει και ένα είδος πλατφόρμα στο Rotterdam όπου συναντιόμαστε και κάθε χρόνο έχουμε ε, μια συνεννόηση για τις ε, χρεώσεις. Ε, Βεβαίω δεν γίνεται σε ατομικό επίπεδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ε, επί τη βάση ε, μιας ε, πολύ επαγγελματικής ετήσιας έκθεσης που είναι μια πάρα πολύ καλή βάση για να συζητηθούν οι χρεώσεις και αν στο τέλος κάποιος έχει κάποιο παράπονο μπορεί βεβαίω πάντα να προσφύγει στα δικαστήρια υπάρχει το δίκαιο του ανταγωνισμού το οποίο κατά την άποψή μας υπερεπαρκεί και ένα σύστημα εποπτείας που θα δημιουργήσει που έχει βεβαίως και την απαραίτητη ε, γραφειοκρατία. Υπάρχει ένα σύστημα ολόκληρο. Και είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το σύστημα, όπως σας είπα, και επηρεάζονται, επηρεάζεται ο ένας από τον άλλον. Οπότε θα ήταν κρίμα με την πρόταση αυτή η οποία αφορά την απελευθέρωση και την εναρμόνιση και τους ίσους όρους ανταγωνισμού. Να καταλήξουμε να έχουμε ε, μια επαναχώρηση και να ρυθμίσουμε κάτι το οποίο δεν χρειάζεται. Συμπέρασμα. Ναι, θέλουμε να σεβαστούμε τις αρχές της συνθήκης, αλλά το ανέφερε και ο ΕΣΠΟ στο έγγραφό του. Δεν θέλουμε να βρεθούμε με έναν κανονιστικό ζουρλομανδία. Δείτε τι γίνεται. Παγκοσμίω με την συγκέντρωση ισχύω αγοράς στα λιμάνια και τονίζουμε την ανάγκη να ενδυναμωθούν τα λιμάνια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος και να παίξουν ένα ρόλο σε μια διεθνή ανταγωνιστική αγορά όπου το Ρότερνταμ βεβαίω ε, ανταγωνίζεται όχι μόνο την Ευρώπη αλλά παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Ε, δεν έχω αντίρρηση να σας δώσω ένα-δυο λεπτά παραπάνω, αλλά όχι και οκτώ, γιατί έτσι στερούμε από τους επόμενους ομιλητές ε, τη δυνατότητα να μιλήσουν όσο χρόνο δικαιούνται. Κύριος Φλάκενστάιν. Αν κατάλαβα καλά, λέτε πως δεν πρέπει να υπάρχει Λέτε πως πρέπει να υπάρχει διαβούλευση και διαδικασίες παραπώνων. Λέτε όμως πως αυτά τα έχουμε και δεν χρειάζεται να τα ξανακάνουμε με κάποια νέα οργάνωση που θα αλλάξει απλά τα ίδια πράγματα. Και έχετε δίκιο πράγματα. Σημαντικό είναι ότι υπάρχει αυτή η διαβούλευση. Σημαντικό είναι να υπάρχει κάπου να απευθυνθεί κανείς και έτσι που τα έχετε οργανωμένα δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταστρέψουμε συστήματα που λειτουργούν. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να το διατυπώσουμε σωστά νομίζω. Γιατί αυτό το οποίο είπατε μου ακούγεται λογικό. Δηλαδή έχουμε ένα τέτοιο σύστημα, δεν χρειάζεται να το καταστρέψουμε και να στήσουμε ένα άλλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά θα περιοριστώ σε τρεις. Ο, η μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι 70% των χρηστών είναι ικανοποιημένοι. Άρα, είναι εύλογο το ερώτημα, είναι απαραίτητη σήμερα η αναθεώρηση με τόσο υψηλό επίπεδο ικανοποίησης. Σε ό,τι αφορά τους παρόχους ε, των υπηρεσιών στα λιμάνια, δεν αναφερθήκατε στο σημείο αυτό. Πιστεύετε ότι η απελευθέρωση της αγοράς και το άνοιγμα στον ανταγωνισμό ανάλογα με τις υπηρεσίες μπορεί να ενοχλήσει, να υπονομεύσει την ποιότητα ή ακόμη και την ασφάλεια στην αυτιλία. Και τι, πού θα γίνει ο διαχωρισμός, στη ρημούλκηση, στην πλοήγηση, στην ε, βυθοκόρηση θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των διαφόρων λιμενικών υπηρεσιών, γιατί για την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα και διατάξεις. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια. Μιλήσατε ε, για μια διάσκεψη που γίνεται συζήτηση για τη χρέωση. Ποιοι συμμετέχουν σε αυτή τη διάσκεψη και πώς γίνεται η συνεννόηση μεταξύ τους για τη χρέωση. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να αυξήσουμε τη διαφάνεια, αν θεωρείτε ότι υπάρχει ε, δυνατότητα για βελτίωση της διαφάνειας, όπως θεωρούμε και εμείς. Και τέλος, για το κανονιστικό επίπεδο, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι ο ρυθμιστικό φορέας που θα πρέπει να πιστοποιεί τι διαδικασίε, Θα πρέπει να είναι εθνικό αυτό ο φορέα, ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκός φορέας ε, ουδέτερος ώστε να μπορεί να λαμβάνει υπόψη τον ε, σεβασμό των κανόνων από όλου του ενδιαφερόμενου. Ευχαριστώ. Άλλο κανεί παρακαλώ. Όχι, έχω κι εγώ μια ερώτηση. Συνεχίζω τι ερωτήσει του κυρίου Σαρίβη. Δεν κατάλαβα ποια είναι η θέση του λιμένου του Ρότερνταμ σε ό,τι αφορά τη ρημούλκηση, τη βυθοκόρηση και την πλοήγηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Σονμέικερ. Σας ευχαριστώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διαβούλευσης και πώς συμμετέχουν οι πελάτες σε αυτήν. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή αυτή η αρχή ε, ότι και ο οργανισμός λιμένος να έχει επαφή με τους πελάτες, ε, γιατί είναι ένας νέος οργανισμός και θα πρέπει να υπάρχει μια πλατφόρμα διαβούλευσης με τους πελάτες. Αλλά είμαστε κατά της υπερβολικής ρύθμισης. Αρκεί να καθορίζουμε την αρχή, ο ορισμός μιας αρχής. Γιατί ο καθένα ε, με διαφορετικό τρόπο χειρίζεται τα πράγματα. Όχι υπερβολική ρύθμιση. Υπάρχει τέτοια πλατφόρμα σε εμά και λειτουργεί θαυμάσια. Τώρα μία επιπλέον παρατήρηση. Εμείς ε, έχουμε ένα διάβλο επαφή με το, μεταξύ του οργανισμού λιμένος και των Χριστών και μάλιστα ε, λέμε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνένεση για τη χρέωση, τότε ανατίθεται ε, το θέμα σε έναν ουδέτερο διαιτητή. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η διάταξη. Είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο σε περίπτωση ασυμφωνίας παραπομπή σε διατησία έχουμε ένα κανονικό σύστημα και για την υποβολή αιτιάσεων και για τις προσφυγές. Κύριε Σουρίμπη, ναι όντως είναι εύλογη η απορία προς τι αναθεώρηση εφόσον το 70% των πελατών δηλώνουν ικανοποιημένοι. Εύλογη ερώτηση, αλλά δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσω. Καλύτερα να την παραπέμψετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η χρηματοδότηση των λιμένων και το πώς ε, ε, θα αξιοποιηθούν οι, οι ευρωπαϊκοί λιμένες προκειμένου να μπουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ε, σε περίπτωση που υπάρχει και κρατική χρηματοδότηση, γιατί εκεί θα δούμε τη διαφορά. Σε ό,τι αφορά τις λιμενικές υπηρεσίες, σίγουρα ο οργανισμός λιμένος εξασφαλίζει ποιότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών. Οπότε η λιμενική αρχή έχει την δυνατότητα να καθορίσει τι εστί καλή και τι κακή ποιότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους. Άρα να υπάρχει διαφάνεια και ορισμός να πληρεί κάποιες προδιαγραφές ποιότητας. Για όλες τις υπηρεσίες του λιμένους. Αλλιώς είναι δύσκολο για έναν οργανισμό λιμένος να διαχειριστεί τα πράγματα με τρόπο που να πληρούνται και οι προδιαγραφές ποιότητας και οι προδιαγραφές ασφάλειας. Κατά τη γνώμη μου δεν θα, υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στην ποιότητα. Γιατί είναι μια άδεια η παραχώρηση που δίνεται από την αρχή του λιμένος στους παρόχους των υπηρεσιών. Οπότε η νέα πρόταση περιλαμβάνει και μια παρατήρηση για την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Το να ε, ξεχωρίζουμε μερικέ είναι πολύ επικίνδυνο ή να εξυπηρετούμε μόνο τους μεγάλους πελάτες και να διαφορούμε για τους ε, μικρότερους. Γιατί κάτι τέτοιο θα έχει αποτέλεσμα την ε, αύξηση των τιμών, των τελών και της χρέας. Κάτι που θα εξοβελήσει τους μικρότερους φορείς. Τώρα, για τη διαφάνεια στη χρέωση. Μιλούμε για τα τέλη στον ιδιωτικό τομέα και για τα τέλη στους λιμένες. Ε, η διαφάνεια στους λιμένες αφορά τη χρέωση των λιμενικών υποδομών. Ε, είπαμε ότι υπάρχει διαδικασία διαβούλευσης και συνένεσης. Σε περίπτωση ε, παραπώνων μπορεί κανείς να προσφύγει στο δικαστήριο ή στην αρχή ανταγωνισμού. Είναι πολύ διαφανής αυτός ο τρόπος για τον καθορισμό των τιμών των τελών και της χρέωσης. Τώρα, για τη χρηματοδότηση μερικές φορές δημιουργεί διαφορετικές τιμές μεταξύ των λιμένων στην Ευρώπη, υπάρχουν κάποια άρθρα στον κανονισμό που μπορούν να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια για να ε, δούμε πώς χρησιμοποιούνται τα κρατικά κονδύλια. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να εξασφαλιστούν συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού. Για να δούμε τι επιτρέπεται από το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τι απαγορεύεται σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των λιμένων γενικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλα τα λιμάνια. Γιατί σε τελική ανάλυση αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα του λιμενικού κλάδου. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε ό,τι, ό,τι εμβαλωματικά μέτρα και να ληφθούν δεν θα αρκούν. Το, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διαφάνεια στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών λιμένων. Θα πρέπει η χρηματοδότηση αυτή να γίνεται όσο πιο διαφάνεια γίνεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, κανονιστική ρυθμίση και αν θα πρέπει να είναι εθνική ή διεθνής, θα ήταν εφιάλτης πραγματικά να ε, υπάρχει κανονιστική ρυθμίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αρκεί η εθνική ρύθμιση. Και πάλι προσοχή. Δεν θα πρέπει να αναχαιτίζεται η εύρυθμη λειτουργία των ήδη λειτουργικών και αποτελεσματικών λιμένων. Σε ό,τι αφορά τους παρόχους υπηρεσιών και ποια είναι η δική μας γνώμη για τις διάφορες υπηρεσίες, κατά τη γνώμη μας η αγορά είναι ελεύθερη, είναι ανοιχτή. Ιδιαίτερα για τα ρήμουλκα και για, τις, για τα για την πλοήγηση, για τους πλοηγούς, η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική, γιατί στο θέμα αυτό υπάρχει ένας, μια ισχυρή πτυχή ασφάλειας. Πιστεύω πάντως ότι όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να ορίζονται με τον ίδιο τρόπο. Στην παρούσα πρόταση είναι υπεραπλουστευμένος ο ε, ορισμός κατά τη γνώμη μου θα πρέπει κάπως να τον προσέξουμε λίγο πιο λεπτομεριακά. Ευχαριστώ κύριε Σολμέικερ. Τώρα πάμε λίγο πιο βόρεια, πιο βόρεια από το Λίβερπουλ, στη Φιλανδία και την Διευθύντρια της Ένωσης Λιμένων της Φιλανδίας, κυρία Ναλίνα Μάκιουλα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε να δείξω ορισμένα ζητήματα όσον αφορά τον προτινόμενο κανονισμό λιμενικών υπηρεσιών. Χαίρομαι που θα μιλήσω μετά τον εκπρόσωπο του λιμανιού του Ρότερνταμ, γιατί εγώ θα μιλήσω για μικρά λιμάνια και για την αγορά των λιμένων αλλά και την όλη βιομηχανική πολιτική. Υπάρχει πολύς ανταγωνισμός μεταξύ των ε, λιμένων και στη Βαλτική θάλασσα συγκεκριμένα με τον ευρύτερο αυτό χώρο και την ε, ευρύτερη αγορά. Ανταγωνισμός γιατί υπάρχουν και λιμάνια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> Μετά το 2015 μάλιστα που θα επιβληθεί η οδηγία για τις εσωτερικές πλωτές οδούς θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Για τον κανονισμό τώρα που συζητούμε. Ο στόχος να αναπτυχθεί η ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σωστός. Η ο χώρος των λιμένων θέλει να παραχθεί ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και στη Φιλανδία, θέλουμε να καλύπτονται περισσότερε υπηρεσίε και να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στου λογαριασμού μα. Θέλουμε ίσου κανόνε ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών λιμένων. Όμω, σε ό,τι αφορά την πρόταση κανονισμού, πρέπει να αναρωτηθούμε εάν τα άρθρα ε, προωθούν ακριβώ αυτό που επιδιώκουμε. Μήπω προκύπτουν μόνο επιχρεώσει για τι λιμενικέ αρχέ, γιατί κατά την άποψή μου θα έπρεπε να υπάρξουν και κίνητρα. Να προσφερθούν κίνητρα για να αναπτύξουν περαιτέρω λιμενικέ αρχέ τι υπηρεσίε που προσφέρουν. Είναι λοιπόν πολύ σωστό το ερώτημα, παρόλο που ξέρω ότι όλη η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα και μακροσκελή. Ο ανταγωνισμό είναι η λέξη κλειδί γιατί η αγορά διαρκώ μεταβάλλεται. Και γι' αυτό νομίζω ότι ο κανονισμός θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ευέλικτος και προσαρμόσιμος. Ε, όσο λιγότερα, τόσο περισσότερα θα αποκομίσουμε. Στην πρόταση αυτή υπάρχουν πολλαπλά άρθρα, τα οποία είναι εξαιρετικά λεπτομερή στη διατύπωση και στις ε, περιγραφές τους. Και ένας λεπτομερέστατος κανονισμός σημαίνει και περίπλοκες διαδικασίες, υποβολή πολλών εκθέσεων και μεγαλύτερο άχθος για τους μικρούς λιμένες. Δηλαδή διοικητικό άχθος στην ουσία. Από τη δική μου την πλευρά το μήνυμα είναι ότι ο κανονισμός θα έπρεπε να είναι ε, ελαφρύς και ευέλικτος. Uh, το πεδίο του κανονισμού νομίζω τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι το κατάλληλο πλαίσιο. Επίσης υπήρξε ένα ερώτημα για τη βυθοκόρηση θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη και από την πλευρά των υποδομών. Θα πρέπει να αποκλείεται νομίζουμε και ε, βεβαίως να δούμε τι θα γίνει επίσης και με, το, με την πλοήγηση στη Φινλανδία. Βλέπουμε ότι η αγορά της πλοήγησης λειτουργεί όλο και περισσότερο και όλο και πιο αποτελεσματικά και γι' αυτό θα θέλαμε να συμπεριλαμβάνεται στον κανονισμό. Όμως, επειδή τα ζητήματα ασφάλειας και προστασίας είναι ευαίσθητα, θα θέλαμε στο άρθρο 6 συγκεκριμένα για σκοπού ασφάλεια και προστασία να περιοριστούν οι παρέχοντε υπηρεσίε και αυτό να συνδυαστεί με το σχέλο τη πλοήγηση. Επίση για του εσωτερικού φορεί, για του εγχώριου φορεί. Να υπάρχει ένα εγχώριο φορέα. Η αρχή διαχείρισης, ο φορέας διαχείρισης θα θέλαμε να είναι ένας και όχι όπως ακριβώς αναφέρεται τώρα στην πρόταση. Τώρα λίγα λόγια για τη Φινλανδία. Και, τις, ε, ξεν, και το εμπόριο με την, ε, και τις εξαγωγές. Το μεγαλύτερο μέρος έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 80% το εμπορικού μας όγκου μεταφέρεται με τις θαλάσσιες οδούς. Όπως βλέπετε όμως στο χάρτη, η Φιλανδία είναι σχεδόν σαν νησί. Είναι μια χώρα με τεράστιες αποστάσεις, αλλά και με μικρές αποστάσεις μεταξύ των λιμένων. Τα λιμάνια μας εξαρτώνται από τις δομές της φιλανδικής βιομηχανίας. Έχουμε κάποιες εταιρείε που είναι παγκόσμια εμβέλειας, όπως η χαρτοβιομηχανία, η βιομηχανία του Χάλιβα και, τον, και η μεταλλουργία και πολλές μικρές ε, βιομηχανίες και εταιρείε, οι οποίες έχουν εργοστάσια ανά χώρα, σε όλη τη χώρα. Οπότε οι κάτοικοι ε, μπορεί να μετακινούνται από τον νότο στο βορρά. Και υπάρχουν λιμένες όλοι όλη μας την αγκογραμμή για το λόγο αυτό. Καθώς και εσωτερικά λιμάνια. Αυτό από την πλευρά της, των λιμένων σημαίνει το εξής. Έχουμε μια δομή με λιμάνια που συνολικά στον αριθμό τους είναι 52, 52 σχετικά μικρά, 10 TNT και 16 μεγάλα. Υπάρχουν πολύ μεγάλος, ε, πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ τους. Τα διευρωπαϊκά λιμάνια καλύπτουν το 19% το 90% μάλλον της εμπορικής κίνησης και το μεγαλύτερο μέρος της επιβατικής κίνησης. 18 εκατομμύρια το χρόνο. Στη Φινλανδία υπάρχουν ε, ένας-δύο μεγάλοι πελάτες ανά λιμάνι, οπότε υπάρχουν λιμάνια όπου υπάρχουν εργοστάσια κοντά στο λιμάνι, ακριβώς δίπλα, που μπορεί να καλύπτουν το 80-90% των εισαγωγών-εξαγωγών ολόκληρου του λιμανιού. Να απασχολούν ολόκληρο το λιμάνι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της Φινλανδίας. Μετά ένα διάγραμμα που ήθελα απλώ να δείτε ότι δεν υπάρχουν μονοπόλια στα φινλανδικά λιμάνια. Είναι κατακαιρματισμένη η αγορά και τα μερίδια της. Έπειτα, τι γίνεται με τα μικρότερα λιμάνια. Απλώς να σας πω ότι τα λιμάνια είναι οργανωμένα τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Τα μικρά λιμάνια μπορούν να είναι επίσης πολύ αποτελεσματικά Και τέλος, τα φιλανδικά λιμάνια θα είναι εταιρείε περιορισμένη ευθύνη από του χρόνου. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει η θεσμολόγηση να γίνεται βάσει τη εμπορική κίνηση. Θα συναντούμε τους πελάτες μας του συναντούμε τόσοι άλλους, του πελάτε και του χρήστε, πολλέ φορέ μέσα στον χρόνο. Δεν χρειαζόμαστε επιτροπή για του ε, χρήστε ξεχωριστή. Και η υποπτική μα αρχή ήδη υπάρχει και υπάρχει και αρχή που διαχειρίζεται τα θέματα ανταγωνισμού. Όπω τα ξέρετε, η Φινλανδία. Μπορείτε να ολοκληρώνετε, παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι, ξέρουμε πολύ καλά τη Φινλανδία, τη γνωρίζουμε. I've even visited the ports of Finland και εγώ επισκέφτηκα και προσωπικά τα λιμάνια της Φιλανδίας και προσπαθώ απεγνωσμένα να τηρήσω το χρόνο και να μην το ξεπεράσουμε γιατί δεν έχουμε για πολλή ώρα την αίθουσα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους 21 νέους από το Βενίτο το Βένετο, συγγνώμη. Χάσατε πριν από λίγο την παρουσίαση του εκπροσώπου του, της οργάνωσης Λιμένος Βενετίας Σας καλωσορίζουμε συνεδρίαση. Κύριε Φλάκινς, αν έχετε ερωτήσεις, ο κύριε Μάισνερ. Αναφερθήκατε κυρία Μέκλερ στο γραφειοκρατικό άκθος που θεσπίζει η πρόταση. Είπατε υπερβολικές α, ε, λεπτομέρειες, πολλές διατυπώσεις, πολλές διαδικασίες. Από εμάς τι περιμένετε, τι θέλετε να διαγράψουμε από τον κανονισμό, ποια σημεία πιστεύετε θα μπορούμε να απαλείψουμε. Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν. Ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ οι οδηγίες υπολογισμού των τελών που πρέπει να είναι ε, NEA εντός Ένωσης. Υπάρχουν κάποια πάγια και κάποια μεταβλητά κόστη ε, που τα υπολογίζετε με βάση την κάθε μεμονωμένη ναυτιλιακή εταιρεία. Γιατί δεν ξέρω, αυτό νομίζω γενικά είναι πολύ, παραπλήσια, πολύ παραπλήσιες χρεώσεις. Τι κάνετε εσείς στην ε, Φιλανδία, κύριε Ζαρβή. Ο κύριος Ζουρίμπη. Ελπίζω ότι θα ολοκληρώνουμε γρήγορα με αυτό το θέμα αυτό. Πολύ σύντομη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σωστά είπατε ότι από τα 1.200 εμπορικά λιμάνια της Ευρώπης, μόνο 328 ανήκουν στα τέντη, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και εμπίπτουν στον κανονισμό. Οπότε από τα 328 αυτά λιμάνια μερικά έχουν 10 πλοία την εβδομάδα, αλλά έχουν χιλιάδες πλοία την εβδομάδα. Πιστεύετε ότι είναι λογικό και συνεπές να έχουμε τον ίδιο κανονισμό που θα επιβάλλεται σε λιμένες που έχουν τόσο διαφορετικά μεγέθη και τόσο διαφορετικό εύρος λιμενικών υπηρεσιών. Λοιπόν, ε, αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι πολύ διαφορετικά τα λιμάνια και τα μεγέθη τους, ε, ενώ ο κανονισμός ισχύει για όλους. Η ερώτηση και του κ. Κουμουτσάκου. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Δεν ξέρω πώς από τα λιμάνια σας ε, λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις. Μπορείτε να μας πείτε. Μπορεί ούτε ένα, αλλά θα ήθελα παρακαλώ απαντήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τώρα θα μιλήσω φιλανδικά. Ευχαριστώ. Κυρία Μάισνερ, σε ό,τι αφορά το γραφειοκρατικό άχθος και τις υπερβολικές διατυπώσεις, το άρθρο 14 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εκεί έχουμε λεπτομέρεια και περιγραφή των διαφόρων διαδικασιών. Υπερβολικά διεξοδική. Αυτό οδηγεί περισσότερο σε αξιολόγηση των επιμέρους διαδικασιών παρά σε υλοποίηση του στόχου. Εγώ θα, προ... θα προτιμούσα μία απλοποίηση του κανονισμού, ώστε να κρατήσουμε τους ίδιους στόχους, αλλά με όχι τόσο ε, διεξοδική περιγραφή της διαδικασίας αναφέρεται κάπου πώς, η Επιτροπή, πώς θα πρέπει να διοργανώνεται η συνεδρίαση της Επιτροπής των Χριστών. Ή τι θα πρέπει, ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο της συζήτησης. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καλύψει μόνο του τα οργανωτικά θέματα. Δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοιο υπερβολικό βαθμό λεπτομέρεια στον κανονισμό. Γι' αυτό μίλησα για γραφειοκρατικό άκθο προηγουμένω και για υπερβολικά λεπτομεριακή περιγραφή των διαδικασιών. Τώρα, αν κατάλαβα καλά τη δεύτερη ερώτηση, μιλήσατε για τη χρέωση. Στην Φιλανδία τα τέλη είναι προσιτά στις διάφορες ιστοσελίδες, μπορεί και κανείς να ενημερωθεί για τις χρεώσεις. Δεν, προσε... δεν προσθέτει τίποτα ο κανονισμός σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει ήδη αρκετή διαφάνεια. Επίσης, θεωρώ ότι ο κανονισμός θα προσθέσει τίποτα σε ό,τι αφορά τη χρέωση. Αναφέρθηκε ε, το μέγεθος των λιμένων. Η διαφορά του μεγέθους. Εμείς έχουμε τρία μεγάλα λιμάνια και 16 λιμάνια μικρότερα που εμπίπτουν όμως στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Εγώ πιστεύω ότι τα λιμάνια που είναι αμυγός εμπορικά μπορούν να είναι αποτελεσματικά άσχετα με το μέγεθός τους. Ακόμη και είναι μικρά, όταν λειτουργούν με εμπορικούς κανόνες μπορεί να είναι αποτελεσματικά. Θα γίνει ένας απολογισμός της κατάστασης, ο συνολικός αριθμός των ε, λιμένων είναι πολύ μεγάλος. Τώρα, για τις κρατικές επιχορηγήσεις. Φέτος ε, είχαμε μερικά λιμάνια που έλαβαν δημοτι... μέχρι φέτος δημοτικές επιχορηγήσεις, αλλά από φέτο θα γίνουν εταιρείε περιορισμένη ευθύνη. οπότε η λειτουργία, η τους θα χρηματοδοτείται από τους πελάτες, από ιδιωτική χρηματοδότηση. Και θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια, γιατί θα ισχύουν μόνο τα εμπορικά κριτήρια και εμπορικοί στόχοι. Σας ευχαριστώ. Ναι, η Φιλανδία είναι πάρα... είναι... έχει σύνορα με την ε, Ρωσική Ομοσπονδία. Με, ακούτε, με καταλαβαίνετε. Η Πετρούπολη, η Αγία Πετρούπολη και το μεγάλο λιμάνι που υπάρχει εκεί πέρα, η, η Λούγκα. Έτσι μιλάμε για κίνηση 120 ε, εκατομμύρια τόνους. Καμία διαφάνεια, τίποτα. Πώς το βλέπετε αυτό από πλευράς ανταγωνισμού. Είμαστε υποδειγματικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, οι άλλοι έχουν άλλο σύστημα εντελώ, έτσι. Σνόντεν ή, Σνόντεν, αυτό συμβαίνει. Βεβαίω, τίθεται και το ζήτημα των παγοθραυστικών επίση, γιατί οι Ρώσοι... Ναι, ναι, το καταλάβαμε, Βέρνερ, ναι, ναι. Τα παγοθραυστικά. Οι Ρώσοι έχουν γίνει πάρα πολύ περιοριστικοί για τη χρήση μη ρωσικών παγοθραυστικών στα ύδατά τους. Μπορείτε να μας απαντήσετε, λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Το λιμάνι αυτό, το Όσλογκα, ε, έχει πράγματι αναπτυχθεί και η κίνησή του είναι ε, η μισή κίνηση όλων των φιλανδικών λιμένων. Και κάποια λιμάνια, ειδικά νότια, έχουν ε, επηρεαστεί πάρα πολύ από τις ε, ροές αυτές, αλλά ο συνολικός όγκος ε, αυτός είναι γύρω στο 7% συνολικά από την Ρωσία δηλαδή, οπότε δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά μας ενδιαφέρει βεβαίως και αυτή η κίνηση και πράγματι τα λιμάνια ανταγωνίζονται μεταξύ τους στη Βαλτική για τα παγωθρευστικά και τη σχέση που έχουν με τον κανονισμό εδώ πέρα. Δεν νομίζω πως ε, έχει τόσο ευρωπαϊκή διάσταση το θέμα αυτό ώστε να συμπεριληφθούν οι υπηρεσίες αυτές ε, στο πεδίο εφαρμογή και δεν νομίζω να έχει προταθεί κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής. Κύριε κύριος Ζανκλωτεριέ, Γενικός Διευθυντής ε, Λιμένος Μασαλίας. Οπότε κατεβήκαμε στα θερμά ύδατα της Μεσογείου από τα παχοθραυστικά. Ζαν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, κυρίες και κύριοι, βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Είμαι πρόεδρος της Διευθυντικής Επιτροπής ε, του λιμένου της Μασαλίας αλλά και της των Λιμενικών Αρχών της Γαλλίας. Γι' αυτό και στις διαφάνειες θα δείτε κάπως ευρύτερες παρατηρήσεις σε σχέση με την απλή περίπτωση της Μασαλίας. Πρώτο στοιχείο, η, γενικές μας, γενική μας αποτίμηση σε σχέση με την πρόταση που μας έχει υποβληθεί. Χαιρετίζω την ε, βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιδιώξει περαιτέρω διαφάνεια και να ε, επαγρυπνεί για την εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών καθώς και να προβλέψει την αυτονομία της διαχείρισης για τις λιμενικές αρχές. Ε, από την άλλη όμως η αντίδρασή μας είναι και μια αντίδραση έκπληξης σε σχέση με το μέσο που έχει επιλέξει, τον κανονισμό, για τρίτη μάλιστα φορά, διότι αυτή τη στιγμή έχει, οι προηγούμενες προσπάθειες έχουν αποκρουστεί ε, και ε, πραγματικά τη χαιρετίζω, την επιμονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μπορεί ένα τέτοιο εργαλείο να καλύψει την πολύ μορφία των διαφορετικών ημενικών πραγματοτικότητων στην Ευρώπη. Η πρόταση, όπως μας έχει υποβληθεί σήμερα, ε, περιλαμβάνει πολύ έντονες αντιφάσεις η πρώτη. Είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη τη συντήρηση. Εδώ πραγματικά είναι πολύ καλή επιλογή αυτή, διότι είναι ένα θέμα εκρηκτικό από κοινωνικής πλευράς και η Μασαλία στο λιμάνι της πλήρωσε ακριβά τώρα τελευταία από την άποψη των συγκρούσεων και κάναμε τα παν για να αποφύγουμε τι εντάσει. Το να υπάρξει ένα κανονισμό για τι λιμενικέ υπηρεσίε και να μην καλύπτεται η βασικότερη υπηρεσία για τα καράβια που είναι η συντήρηση είναι εκπληκτικό. Επίση, μιλά για την αυτονομία των λιμενικών αρχών η πρόταση τη Επιτροπή, αλλά προσπαθεί να πλαισιώσει με πολύ δεσμευτικό και περιοριστικό τρόπο ε, τι κινήσει του. Κατά τρίτον, θεωρούμε ότι κάπω διαστρεβλώνει την αρχή τη επικουρικότητα που επαναλαμβάνω εξορισμού μα φαίνεται ότι θα μπορούσε να καλύπτει καλύτερα την ποικιλομορφία των ε, διαφορετικών πραγματικότητων στα λιμανιά τη Ευρώπη. Άρα, σε πρώτη φάση, η αντίδρασή μα είναι απορριπτική. Τίνουμε να απορρίπτουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που μοιάζει με ένα πυρηνικό όπλο η απόρριψη, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκρηκτικέ ε, και αλυσιδωτέ αντιδράσεις. Πάντω, εάν το Κοινοβούλιο συνεχίσει να προωθεί την εξέταση τη πρόταση αυτή του κανονισμού, ε, θα υποβληθούν πολυάρεθμε τροπολογίε προκειμένου να βελτιωθεί σε σχέση με τη σημερινή τη παρουσίαση πρόταση. Πρόεδρε, να περάσω τώρα σε πιο συγκεκριμένε παρατηρήσει ε, και σε ερωτήματα που ενδεχομένω σα απασχολούν. Πρώτον, το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Πιστεύουμε ότι η βυθοκόρηση θα πρέπει να αποκλειστεί, διότι μιλάμε για την συντηρήση των λιμενικών υπηρεσιών μεν, αλλά δεν είναι μια υπηρεσία που να προσφέρεται για τα καράβια αυτή για τα πλοία. Επίσης, το άρθρο 9. Νομίζουμε ότι περιπλέκει τα πράγματα εφόσον απαιτεί να γίνεται διασύνδεση μεταξύ του ελέγχου και της παρακολούθησης της από την αρχή που αποφασίζει για τις δημόσιες υπηρεσίες και του φορέα που προσφέρει τις υπηρεσίες στην αγορά. Αυτό μας φαίνεται εξαιρετικά περιοριστικό έτσι όπως ε, εκφράζεται και δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις πραγματικότητες που συναντούμε ανά την Ευρώπη. Ως προς τους παρέχοντε υπηρεσίε. Θα μπορούσε ένας ιδιωτικό φορέας να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες. Εφόσον υπάρχει έλεγχος, αυτό καλύπτεται. Αλλά δεν ανάγκη να υπάρχει τόσο αυστηρή ιεράρχηση ω προ την ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων διαφάνεια και της εμπορικής, του ελεύθερου εμπορίου, είναι νομίζω απλά τα πράγματα. Το λιμάνι τη Μασαλία υπόκειται στου κανόνε τη ε, οδηγία για τη διαφάνεια. Δεν βρίσκουμε το λόγο να πάμε πιο μακριά σήμερα. Γιατί χρειάζεται περαιτέρω ε, ρύθμιση για τα λιμάνια. Και ακόμα και αν το θέμα αυτό παραμείνει, τουλάχιστον να περιοριστεί στι υπηρεσίε για τι οποίε ο υπεύθυνο για τη διαχείριση έχει δημόσια χρηματοδότηση. Δεν το έχουμε πει νομίζω επανειλημμένω. Πρέπει να το ξαναπούμε ακόμη και να ακούστηκε ότι θέλουμε να έχουμε ανοιχτή και ελεύθερη αγορά. Ωραία. Αλλά δεν βλέπουμε την ανάγκη να ε, διαλύσουμε τη διαμόρφωση του κόστους και των τιμών, μάλλον να τι αναλύσουμε τόσο εξονυχιστικά, ενώ υπάρχουν υποχρεώσει υποβολή εκθέσεων και πληροφοριών και για το επίπεδο των τιμών και για τι διακυμάνσει του, αλλά και για την ε, πολιτική μα ως προς τι τιμέ και από μακροοικονομική προοπτική σε σχέση με την κατάσταση τη αγορά, τι επενδύσει που γίνονται, ε, το benchmarking, όλα αυτά δίνουν κάποιου γενικού ε, προσανατολισμούς. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τα ε, ξεπεράσουμε ω προ τα ιδιωτικά λιμανιά. Θα συμφωνήσω με την άποψη του προσώπου του λιμανιού του Ρότερνταμ. Δεν θα πρέπει να τα αποκλείσουμε, διότι θα υπήρχε στρέβλωση του ανταγωνισμού και αν πρέπει να βρούμε μια κοινή γραμμή, θα έπρεπε να αναζητήσουμε ως κριτήριο το μέγεθος των λιμένων. Και από εκεί να δούμε τι θα συμπεριληφθεί και τι θα αποκλειστεί. Η οδηγία ε, για τη διαφάνεια έχει ως όρο τα 49 εκατομμύρια τόνους. Ε, και έπειτα για την αρχή του ελέγχου, στη Γαλλία υπάρχουν συστήματα, έχουμε αρχή υπεύθυνη για τον ανταγωνισμό, για τα θέματα ανταγωνισμού, που κάνει πολύ προσεκτικές επιλογές. Έχουμε το ελεκτικό συνέδριο που ασχολείται με τα μεγάλα λιμάνια και τις εμπορικές τους κινήσεις και όχι μόνο με τους λογαριασμούς τους, αλλά και το πώς αξιοποιούνται τα δημόσια κονδύλια και κάνει και συστάσεις. Έχουμε επίσης δικαστήρια. Όλα αυτά ε, λειτουργούν μια χαρά, λειτουργούν εύρυθμα, υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Δεν βλέπουμε την ανάγκη να υπάρξει περαιτέρω διαστρωμάτωση. Τέλος, για να ολοκληρώσω, δεν πρέπει να υπερεύσει το χρόνο μου παρά μόνο κατά δύο λεπτά, ως προς τις δεσμεύσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν νέα θέματα για τα λιμάνια, όπως οι ανταποκρίσει για τι οποίε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα τα λιμάνια όπω αυτό τη Μασαλία, αλλά θα πρέπει να πλουστεύσουμε εδώ τι διαδικασίε. Δηλαδή να ενισχύσουν, να ενισχύσουν τι επιδόσει του τα λιμένε αλλά και να δούμε πώς μπορεί να υπάρχουν καλύτερες υπηρεσίες χερσαίες. νομίζω ότι αυτό είναι καθοριστική σημασία για τα λιμάνια. Νομίζω παρέμεινα σε ένα τρίλεπτο υπέρβαση του χρόνου μου, Πρόεδρε, όπως μου είχατε επιτρέψει. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Φλέκενστάιν. Μία σύντομη ερώτηση έχω μόνο για τις χρεώσεις τέλη. Μπορείτε να μας πείτε πού θα βάζατε εσείς τη, τη γραμμή, το όριο. Ίσως να μην σας κατάλαβα καλά. Γιατί πρέπει να είναι δεσμευτικό και τι όχι. Δηλαδή. Ευχαριστώ κύριε Βουέλς. Ευχαριστώ. Κύριε Τεριέ, θεωρείτε πως είναι καν απαραίτητος ο κανονισμός. Στη μελέτη ήταν 80% ικανοποιημένοι με την αγορά που επικράτει και κάποιοι άλλοι βλέπουν μεγαλύτερο ρόλο των ναυτιλιακών εταιριών το οποίο, θα, το οποίο θεωρούν πρόβλημα. Τι άποψη έχετε, ο κύριος Κουμουτσάκος. Ε, κύριε Τεργέ, δεν ε, κατανόησα στην αρχή της παρεμβάσεώς σας Κατάλαβα ότι θεωρείτε ότι μια τρίτη προσπάθεια από πλευράς Επιτροπής να έρθει ένας νέος κανονισμός ε, για σας είναι ακατανόητη. Δεν θέλετε τίποτα ή θέλετε ένα άλλο κείμενο, ας πούμε μια οδηγία ή κάτι άλλο. Ο κανονισμός είναι που ενοχλεί ή δεν θέλετε καμία προσπάθεια από πλευράς Επιτροπής. Κύριε εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στις υπηρεσίες. Ε, ο κύριος Τεργέ είπε θα προτιμούσε η βυθοκόρηση να αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Γιατί έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η βυθοκόρηση. Είναι περισσότερο θέμα συντήρηση υποδομών. Αλλά τι γίνεται με τη ρημούλκηση, με την πρόσδεση, με την πλοήγηση. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ αυτών των ε, υπηρεσιών. Ε, στο όνομα της ασφάλειας ε, των μεταφορών. Για τους πλοηγούς πιστεύω ότι θα πρέπει να τους ε, αποκλείσουμε από το πεδίο εφαρμογή. Γιατί στη Γαλλία υπάρχει ένα σύστημα συνεταιριστικό που προϋποθέτει πολύ σημαντικές επενδύσεις. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνουμε ανοιχτούς διαγωνισμούς προς όλες τις κατευθύνσεις ή να αφαιρέσουμε τους πλοηγούς από το, από το πεδίο εφαρμογή τους από το πεδίο του κανονισμού. Σε ό,τι αφορά το, την ενεργειακή μετάβαση. Ποιος είναι ο ρόλος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί και βολονταριστικοί απέναντι στους ευρωπαϊκούς λιμένες. Γιατί έχει, έχουν ε, πτυχή εμπορική, αλλά έχουν και κοινωνική πτυχή οι λιμένες. Πιστεύετε ότι και αυτή η πτυχή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Κύριε Τεριά, παρακαλώ. Δεν είμαι ε, σίγουρος ε, για την διευκρινιστική ερώτηση που μου έκανε ο εισηγητής ως προς τις χρεώσεις. Τι θέλετε ακριβώς να διευκρινίσω κύριε εισηγητά. Κνούτ, μπορείς να επαναλάβεις την ερώτησή σου. Υπενθύμησέ μας ακριβώς τη ρώτησες. Πού βρίσκομαι κύριε Πρόεδρε. Πού βρίσκομαι. Λοιπόν, ε, ήθελα να μάθω στο θέμα της διαφάνειας στη διαμόρφωση των τιμών που ε, βάζετε εσείς τη γραμμή τι πρέπει να είναι υποχρεωτικά διάφανο και που λέτε, εντάξει, σταματάει η πλάκα, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε τα ε, συμφέροντα της εταιρεία που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Κύριε Εταιρεία. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο είναι να αναλύσουμε πλήρως ε, τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε το κόστος ε, και τις ε, τιμές, τα τέλη. Βέβαια, όταν λαμβάνουμε δημόσιες επιδοτήσεις, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία, αναφυσβήτητα. Εμείς ως ελεύθεροι φορείς διαχείρισης θα πρέπει να έχουμε την εμπορική αυτή ελευθερία, να μην χρειάζεται να τα, υπολογίσουμε, να τα εξηγήσουμε όλα με την παραμικρή λεπτομέρεια στους πελάτες. Από τη στιγμή που σε προηγούμενο στάδιο έχουμε διαβούλευση μαζί τους για την πολιτική των τελών, αλλά άλλο διαβούλευση για την πολιτική των τελών και άλλο για το ύψος των τελών. Υπάρχει διαχωρισμός εδώ. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ερώτηση. Η οδηγία για τη διαφάνεια και η οδηγία για τις παραχωρήσεις καλύπτουν ε, τις, ε, όλες μας τις ανησυχίες. Η αναγκαιότητα ενός κανονισμού δεν είναι αυτονόητη εδώ. Και όταν ε, μίλησα προηγουμένως για το θέμα αυτό, αναφέρθηκα στις προηγούμενες απόπειρες που έγιναν. Είπα ότι είναι η τρίτη ήδη απόπειρα αυτή. Οπότε, ως Ω προ τον κανονισμό, ακούστηκε επίκριση ότι είναι σα βουρλομανδία, υπερβολικά ασφικτικό κλειό, είναι υπερβολικά δεσμευτικό. Και η τελευταία εκδοχή, κατά τη γνώμη μου, είναι ακόμη πιο περιοριστική, αν επιμείνουμε σε αυτή την ιδέα του κανονισμού. Εγώ δεν είπα ότι αρνούμαστε την αρχή, αρνούμαστε τον κανονισμό, αλλά θα πρέπει να ενταχθούμε σε μια θετική δυναμική για να προωθήσουμε και το κανονιστικό πλαίσιο. Πάντως πιστεύουμε ότι οι οδηγίες είναι πολύ καλύτερα νομοθετικά όργανα και ότι υπάρχουσες οδηγίες καλύπτουν εκτενώς τις ανησυχίες μας και τα προβλήματα, τους προβληματισμούς. Κύριε Ζουριμπή, δεν θα επανέλθω στο θέμα της βυθοκόρησης. Τώρα το θέμα της πλοήγησης. Ε, είναι δικαιολογημένο και αποδοτικό το σύστημα, γιατί καλύπτονται και οι πτυχές της ε, ασφάλειας και θα πρέπει φυσικά να λαμβάνονται υπόψη ανα πάσα στιγμή. Για άλλες υπηρεσίες τώρα, ίσως το μέγεθος της αγοράς ε, μπορεί να δώσει δουλειά σε έναν πάροχο και αν είναι πολύ μικρή δουλειά να, να μην επιβιώνουν. Θα πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν εχέγγυα για, τις, ε, για τα τέλη. ό,τι αφορά τη ρημούλκηση, έχουμε ένα σύστημα που μιλάει για έναν ελάχιστο αριθμό κοιτών που θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για να μπορεί ε, να ρημουλκίσει ένα μεγάλο δεξαμενόπλιο, ειδικά σε αντίξωες καιρικές συνθήκες. Οπότε δεν θα πρέπει να δημιουργούμε εμπόδια για την είσοδο ε, στην αγορά νέων παρόχων, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πάνω από όλα τις πτυχές της ασφάλειας και πρώτα αυτό να εξασφαλίζουμε και ως προς την ρημούλκηση. Τώρα, για το κατά πόσο ε, λαμβάνεται υπόψη μόνο το θέμα το εμπορικό και όχι το θέμα το χωροταξικό, που επίσης είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά τους λιμένες. Έχουμε όμως την οδηγία για τις παραχωρήσεις, που περιλαμβάνει και κάποιες τέτοιες προοπτικές. Πάντως και η χωροταξική διάσταση του λιμένων είναι πολύ σημαντική. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ενεργειακό ζήτημα, ο λιμένας της Μασαλίας ε, την τελευταία πενταετία ε, βίωσε μία μίνι πετρελαϊκή κρίση με τις συνέπειες για, τις, για τα ευρωπαϊκά δηληστήρια και ουσιαστικά φτιάχνουμε τώρα ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Και σίγουρα εκεί θα χρειαστούμε πολλές πρωτοβουλίες και ένα πολύ αίσιο κλίμα που θα δημιουργήσει η Ευρώπη, ελπίζουμε, στο τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Now it's, um, we go on to... ευχαριστώ, κύριε Τεριέ. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πέντε λεπτά. Ποιος θα μιλήσει. Πέντε λεπτά έχετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους των λιμένων που μοιράστηκαν μαζί, τους, μαζί μας την σοφία τους. Απόψε δεν φιλοδοξώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω κάποια πράγματα. Η Κομισιόν την διαβούλευση την ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια, από το 1997 τουλάχιστον, στη συγκεκριμένη πρόταση από το 2011. Όσοι είναι στο κορυφαίο επίπεδο ξέρουν πόσες φορές έχουμε συναντηθεί, οπότε δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς για έλλειψη διαβούλευσης. Μπορείτε να μας πείτε γιατί το χρειαζόμαστε, τα λιμάνια λειτουργούν. Ε, Μιλήσετε για νούμερα όπως 70%. Να σας πενθυμίσω πως σε κάποιες υπηρεσίες τα νούμερα είναι κάτω από 50% ικανοποίηση χρηστών. Επίσης, σύμφωνα με τις μελέτες του ΟΣΑ, 40% των ευρωπαϊκών λιμενικών υποδομών είναι κάτω του μετρίου παγκοσμίω. Όσον αφορά δε την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας ε, υπάρχουν ε, ευρωπαϊκές χώρες που είναι στην 76η θέση από τις 100. Ε, κατά μέσο όρο πάμε καλά, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε καλά σε όλα τα λιμάνια. Αυτή πρέπει να είναι η φιλοδοξία μας. Επίσης, ο όρος Ζουρλομανδίας είναι και μη αναλογικός και λανθασμένος από όσους βρίσκονται εδώ πέρα, ιδιαίτερα τους ε, βουλευτές, ε, έχετε δει πως είναι οι κανονισμοί της αεροπορίας, του σιτηροδρόμου, των οδικών μεταφορών και οι κανονισμοί ε, της ναυτιλίας, όπου έχουμε δεκάδες κανονισμούς, έτσι, δεκάδες σελίδες ονομάτων κανονισμού. Εδώ πέρα η πρόταση η οποία ε, περιέχει απλά τα βασικά της συνθήκης, δηλαδή την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και την αρχή της διαφάνειας, ε, δεν το λες και ζουρλομανδία, είναι κάποια εργαλεία τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν σε ε, όλες τις καταστάσεις. Και σας προκαλώ να μου δώσετε ένα παράδειγμα όπου το οργανωτικό σύστημα του λιμανιού κάνει ε, διαφορά στι πολύ βασικές αρχές που ανακοινώνουμε εδώ πέρα με τον κανονισμό αυτόν. Κάποια άλλα λεπτομεριακά ζητήματα. Μιλήσατε για κρατικέ ενισχύσει, ανάπτυξη λιμένων, διαφάνεια. Χαίρομαι για το ότι όλοι συμφωνείτε. Επίσης, μιλήσατε για ζητήματα όπως το ότι κάποιες υπηρεσίες πρέπει να συμπεριληφθούν ε, όπως ε, η πλογή. Ποιο είναι το θέμα, ασφάλεια, ανεξαρτησία και να μην διαλέγει κανείς μόνο αυτά που θέλει. Ε, το νομίζαμε το είχαμε καλύψει. Αν δεν επαρκεί, ευχαρίστω να συνεργαστούμε μαζί σας για να ξεκαθαρίσουμε πώς. Εμείς πιο πολύ από όλα τα άλλα όργανα δεν θέλουμε να πέσουν ε, οι προδιαγραφές ασφαλείας. Ε, τα φτιάχνουμε εδώ και δεκαετίες, δεν θέλουμε να χαμηλώσουν τώρα. Όσον αφορά το διοικητικό βάρος και τη γραφειοκρατία, βλέπετε δεν υπάρχουν υποχρεώσεις αναφοράς, τα δεδομένα θα είναι στην διάθεση ε, αυτών που μπορούν να τα εξετάσουν. Θα δείτε πως δεν υπάρχουν νέες δομές που ζητάμε να δημιουργηθούν και εδώ πέρα συμφωνώ πλήρω με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φλέκενστάιν, δηλαδή αν είναι να παραπονεθεί, να υπάρχει κάπου να παραπονεθεί κανείς, είναι καλό. Αν μου λέτε το έχουμε, τι το θέμε, Α, δεν χρειάζεται. Το έχετε, τελείωσε. πατήστε τσικ στο κουμπάκι και τελείωσε. Ίσως άλλοι να μην έχουν τέτοια υπηρεσία που είναι στο 40% των λιμένων της Ευρώπης που δεν, είναι, δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά. Ε, σημαίνει πως υπάρχει όμως ουσιαστικός λόγος για να δημιουργηθεί κάτι. Κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα, στις αίθουσες αυτές εδώ μέσα ε, διαπραγματευτήκατε το νέο διευρωπαϊκό δίκτυο, κάτι το οποίο χρειάστηκε 30 χρόνια να οριστικοποιηθεί, το οποίο βασίζεται στους βασικούς κανόνες της διαφάνειας, ε, δίκαιης πρόσβασης στην αγορά, ασφάλεια και διαλειτουργικότητα. Οπωσδήποτε δεν θα πείτε πως τώρα όσον αφορά τα λιμάνια δεν χρειαζόμαστε αυτές τις αρχές. Αντιθέτως, αυτό το οποίο θέλουμε είναι εσείς να μας βοηθήσετε έτσι ώστε οι βασικές αυτές αρχές που υπρασπίζετε τα τελευταία χρόνια να συνεχίσουν να ισχύουν και για το ευρωπαϊκό λιμενικό σύστημα, τις πύλες μας στον κόσμο και Βεβαίω ε, τους κινητήρες της ανάπτυξης ε, στην Ευρώπη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στις καταληκτήριες παρατηρήσεις του εισηγητή και Πρόεδρου. Ο εισηγητής πρόεδρος ο κ. Φλακοστάνη. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όσους μας βοήθησαν σήμερα με τις παρουσιάσεις τους δεν θα αναφερθώ σε όλα τα θέματα, δεν είναι αυτή η δουλειά μου σήμερα. Ακούσαμε πως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το σε ποιο βαθμό πρέπει να συμπεριληφθούν τα ιδιωτικά λιμάνια στον κανονισμό ή όχι. Ακούσαμε πως πρέπει να δούμε πάρα πολύ προσεκτικά τι γίνεται με τις χρεώσεις, το τι είναι διαφάνεια και που ξεπερνάμε το όριο και βλάπτουμε την εμπορική πολιτική του κάθε λιμένα. Θέλω να πω κάτι ακόμα το οποίο δεν αναφέραμε. Οι πράξεις κατεψιοδότηση εδώ πέρα πρέπει να περιοριστούν στο απολύτως ελάχιστο. Κάτι άλλο δεν αναφέραμε σήμερα γιατί ίσως να μην είναι τόσο σημαντικό για τα λιμάνια, αλλά ενισχύεται η αυτονομία των λιμανιών μέσω αυτού του κανονισμού και αυτό το θεωρώ σημαντικό και αυτά τα οποία εγώ ε, επισκέφτηκα εκεί όπου καθορίζονται τα τέλη στην πρωτεύουσα και όχι στο λιμάνι νομίζω θα χαρούν. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, άκουσα πως ε, βυθοκόροι δεν ε, εντάσσονται γιατί δεν ανήκουν σε αυτό. Έχουμε αρκετά να κάνουμε σε αυτό ακόμα. Ε, για τους δε πλοηγούς, επειδή είναι ζήτημα ασφάλειας, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια. Η πρόσβαση στην αγορά είναι κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ επίσης για το ότι έχουν μείνει εκτός οι επιβάτες και τα εμπορεύματα. Ξέρω πως οι ναυτιλιακές εταιρείε που δεν βρίσκονται εδώ πέρα σήμερα τα βλέπουν ε, ε, διαφορετικά, αλλά θα πρέπει να έρθουμε και σε επαφή μαζί τους. Σημαντικό είναι δούμε τον ε, αριθμό των ε, ανταγωνιζομένων. Πρέπει να υπάρχει και μια οικονομική λογική. Σε ένα μικρό λιμάνι δεν μπορεί να είναι δίπλα-δίπλα δύο ανταγωνιστές όταν υπάρχει δουλειά ίσα-ίσα για έναν. Πρέπει να δούμε έναν τρόπο να το διατυπώσουμε λογικά όμως αυτό. Για το δικαίωμα διαβούλευσης των χρηστών και αυτό το οποίο ε, για το, τη, τον καθορισμό της Κομισιόν ως ε, φορέα διαβούλευσης. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά η αρχική σας πρόθεση είναι πως δεν μπορούμε να πούμε ένα σύστημα για όλους. Μιλήσατε για κάποια εργαλεία, ε, αλλά πρέπει να το γράψουμε εδώ πέρα πιο ξεκάθαρα, έτσι ώστε το πρόβλημα το οποίο αναφέρατε να λυθεί κιόλας να πω επίσης κάτι για το μέλλον. Πρώτον, ο κανονισμός δεν μπορεί να ειδωθεί σε ένα κενό, αν θέλετε. Πρέπει να κριθεί και να αποφασιστεί μαζί με την οδηγία περί συμβάσεων παραχώρησης, γιατί σχετίζονται πάρα πολύ στενά. Έχει υπάρξει. Αν ε, υπάρξει λοιπόν συμφωνία και για την αλληλοδηγία στις άλλες επιτροπές των αρμόδιες, ελπίζω να τα καταφέρουμε και εμείς. Και κατόπιν τα έγγραφα για τις κρατικές ενισχύσεις που περιμένουμε ε, αρχή του επομένου έτους, νομίζω θα μας βοηθήσουν. Νομίζω δεν είναι από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, αλλά από τη Γενική Διεύθυνση του Ορθού Λόγου, του ανταγωνισμού δηλαδή. Τέλος Νοεμβρίου Αναμένουμε την έκθεση η οποία θα, αποτελείται από θα έχει 84-85 τροπολογίες. Αναμένουμε ακόμα τη μετάφραση βεβαίως από τα αγγλικά. Ελπίζω να μπορέσουμε να συναντηθούμε. Αλλά δεν υπάρχει νομίζω αρκετός χρόνος μέχρι τέλος Δεκεμβρίου αρχές Ιανουαρίου πρέπει να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε για να μπορέσουμε να έχουμε στο τέλος κάτι που θα είναι αντικείμενο νομίζω συμφωνίες για την προσθέμενη αξία κάτι αναφέρθηκε τώρα στις επισκέψεις μου σε διάφορα λιμάνια άκουσα τους ε, περισσότερους ε, ενδιαφερόμενους που μου είπαν εντάξει θα γίνουν κάποιες διορθώσεις και θα τελειώσει αυτή η συζήτηση και για λίγα χρόνια θα έχουν λίγο την ησυχία τους. Αυτό θέλω ως αποτέλεσμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια σας. Thank you, Mr. Fleckenstein. Ευχαριστούμε κύριε Φλέκενστάιν. Εγώ επιβεβαίωνω ότι ελπίζουμε στις 26 Νοεμβρίου να έχουμε το σχέδιο έκθεσης για εξέταση και τότε θα ορίσουμε και μια προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Θα έχουμε δηλαδή τουλάχιστον δύο ακόμη συζητήσει στην Επιτροπή Μεταφορών πριν την ψηφοφορία. Ο κύριος Φλακεστάιν πάντως έχει αρκετά δύσκολο έργο και το πρώτο βασικό ερώτημα είναι είναι τροποποιήσιμη αυτή η πρόταση έχετε βελτιώσεις. Ή μήπως θα πρέπει να την απορρίψουμε όλος χερός. Από αυτή την άποψη είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι αν αφαιρέσουμε τη διακίνηση φορτίου και από ό,τι κατάλαβα από τα κράτη-μέλη, αν αφαιρέσουμε και την πλόγηση, αν αφαιρέσουμε και την βυθοκόρηση, τότε τι θα μείνει στον κανονισμό. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί λοιπόν καλά ο εισηγητής και να υποβάλει πρόταση στην Επιτροπή για το ποια είναι η γνώμη του και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως από τις σημερινές ομιλίες και παρουσιάσεις και από τις ερωτήσεις που έγιναν, έχουμε ήδη ένα καλό σημείο αφετηρίας και αρχίζουμε σιγά σιγά και κατανοούμε καλύτερα αυτόν τον κλάδο των μεταφορών. Άκουσα και τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι ο κανονισμός για τους σιδηροδρόμους είναι ότι καλύτερο είχαμε στην ε, κοινοτική νομοθεσία. Παρά κάποια επιτέγματα τώρα, σε ό,τι αφορά τις προτάσεις ε, για την ε, αεροπορία, ιδιαίτερα οι προτάσεις για, τους, για τα αεροδρόμια η πρόταση έχει κολλήσει στο Συμβούλιο. Από εκεί είναι που κινητοποιηθήκαμε. Μας το λέτε ως παράδειγμα για πρόοδο λοιπόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις οδικές μεταφορές, σήμερα το πρωί είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση για τις οδικές μεταφορές. Και φαίνεται ότι πολλοί ούτε και αυτό το θέμα το θεωρούν καταπληκτικό. Θα δούμε όμως τι θα βγει τις επόμενες εβδομάδες από τις συζητήσεις. Ευχαριστώ πάντω τον Ζαν Κλοντ Τεριέ από το λιμένα τη Μασαλία, την Αναλίνα Μάκουλα από τα Φιλανδικά λιμάνια, τον Βίκτορ Σον Μάκερ από το λιμένα του Ρότερνταμ, τον κύριο Στεφάνο Μπενάλντο από τον Οργανισμό Λιμένος Βενετίας και τον Ρίτσαρντ Μπέρτ από την Ένωση Μιζώνων Λιμένων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους και ευχαριστώ θερμά και τους ευρωβουλευτές για τη συμμετοχή τους στη συζήτηση και μπορούμε πια να πούμε ότι περιμένουμε με αδημονία και ενδιαφέρον το σχέδιο έκθεση του κ. Φλάκενστάιν. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η μήνυα κρόαση.